Τέσσερα λεπτά στην κυρία Βάτμαντς. Και μετά θα περάσουμε στο Κατσιάι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν να διασφαλίσουμε καλύτερα την ασφαλεία τους. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφέ ότι χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ναι, αλλά και μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε όλους τους κλάδους. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός ε, τομέας ε, ε, λειτουργούν, συνεργάζονται μάλλον ανεπαρκώς αυτή τη στιγμή. 3,5 εκατομμύρια πολίτες, 1,5 εξ 1,5 εκατομμύρια από αυτού στην Ευρώπη εργάζονται σε εταιρείε ιδιωτική ασφαλεία. Ε, όμως ε, δεν, υπάρχει δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για τη λειτουργία αυτών των εταιρείων ασφαλείας. Χρειάζονται ε, συγκεκριμένα πρότυπα εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών, παρακολούθηση της λειτουργίας τους και να εξασφαλίσουμε ένα κοινό νομικό πλαίσιο για το χειρισμό των δεδομένων. Χρειαζόμαστε λοιπόν από την ε, Κομισιόν μια οδηγία έτσι ώστε να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και να αποκτήσουμε κοινού κανόνες για όλες αυτές τις ιδιωτικές εταιρείε ασφαλείας. Θα πρέπει να καταγράψουμε όλες τις εταιρείε που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαθέτουμε, επαναλαμβάνω, κοινού κανόνες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιωτικές εταιρείε ασφαλείας χρησιμοποιούνται και εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάρο τη εικόνα που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα λοιπόν το πώς λειτουργούν, διότι ε, πολύ συχνά οι δραστηριότητες τους ξεφεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνουν μέχρι και τη χρήση όπλων. Η έκθεση αυτή είναι αρκετά φιλόδοξη, κάνει, απευθύνει αρκετέ συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι θα τι λάβει υπόψη τη. Μία από αυτέ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, ζητούμε από την Κομισιόν να υποβάλει μια πράσινη βίβλο. Γνωρίζω ότι υποβάλλονται πολλέ πράσινε, λευκέ και άλλων χρωμάτων βίβλοι, αλλά χρειαζόμαστε μια πράσινη βίβλο που, στην οποία θα συνεισφέρουν ε, όλοι οι φορεί ιδιωτικού και δημόσιου κλάδου που εμπλέκονται στον ε, τομέα αυτό και θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και κύριε Μογκερίνη, αυτό χρειάζεται διότι με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση, το πανόραμα και θα αποφύγουμε ε, τις ε, καταχρήσεις ε, οι οποίες παρατηρούνται στον τομέα χρειαζόμαστε περισσότερη άμυνα με λιγότερα χρήματα, γίνονται περικοπές στον ε, αμυντικό προπολογισμό ε, σε όλα τα κράτη-μέλη, χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα και ο πειρασμός είναι να ε, δίνουμε υπεργολαβία αυτά τα καθήκοντα σε τέτοιου είδου εταιρείε. Δεν μπορούμε όμως αυτές οι εταιρείε να τις αφήσουμε χωρίς έλεγχο. Μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε μόνο αν διαθέτουμε τους κατάλληλους κανόνες ε, επιτήρησης τους. Ε, θέλω να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να σας ζητήσουμε ε, να υποβάλλετε μια, ένα προσχέδιο οδηγίας και κάποιου προσωρινούς κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίσουν την δημιουργία και τη λειτουργία εταιριών ιδιωτικής ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να υποκαθιστούν στρατούς χωρίς να έχουν συγκεκριμένους κανόνες. Δεν δεν είναι δυνατόν επίσης ε, να ε, ε, επεκτείνουν τις δραστηριότητε τους σε στρατιωτικά καθήκοντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που με βοήθησαν και ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια που τηρήσατε και το χρονικό όριο για την ομιλία σας και για την παρέμβαση καθ' αυτή. Τώρα, catch the eye, πέντε λεπτά, ο κύριος και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είπατε εκπρόσωπε, αναγνωρίζω ότι ως ένα βαθμό περιορισμένο αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας μπορεί να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αμυντικά καθήκοντα, αλλά δεν συμφωνώ με την έκκλησή σας να εγκρίνουμε νέες οδηγίες διότι πιστεύω ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ε, συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουν αυτοί περισσότερα δικαιώματα από τον απλό πολίτη. Νομίζω ότι η ανάθεση σε ε, τέτοιες ε, εταιρείε όπως περιγράφει η εισηγήτρια είναι αρνητική εξέλιξη και θα πρέπει να θεσπίσουμε τις κατάλληλες συστάσεις που θα τις στηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Κατερίνα Καμίτσι. Ε, Signora Alto Rappresentante, negli ultimi anni il settore della sicurezza privata effettivamente ha conosciuto una forte espansione. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στους προϋπολογισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Η εξωτερική ανάθεση σε τέτοιες εταιρείες κατέστη επιτακτική. Ε, πρέπει να ελέγχουμε τις διαδικασίες ε, και να φροντίζουμε να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν και αυτές πηγαίνουν πέρα από την ανάγκη περιορισμού του κόστους. Χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμός ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά θέματα, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και τα επιχειρησιακά. Ε, θα φροντίσουμε λοιπόν οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας θα λειτουργούν σωστά ιδιαίτερα όταν ε, λειτουργούν σε τρίτες χώρες και θα έχουμε ευθύνη να επισημαίνουμε τις... Ε, θα σας ευχαριστούμε κύριε Κινίτσο, κύριο Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το συνταγματικό δίκαιο και η πολιτική επιστήμη γνωρίζουμε ότι καθορίζουν ότι το κράτος έχει το μονοπόλιο της άσκησης της νόμιμης βίας. γι' αυτό και η άμυνα και η ασφάλεια ανατίθεται σε δημόσιες αρχές. λόγω του νεοφιλελευθερισμού αυτό που βλέπουμε είναι πλέον να ανατεθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να ασκούν βία και μάλιστα αυτή να θεωρείται και νομιμοποιημένη. αυτό είναι ένα παράδεκτο φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί είδαμε αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν και στο ιράκ και άσκησαν και στρατιωτική δράση. είδαμε εταιρείες τέτοιες να κατηγορούνται για βασανιστήρια για απώλεια ζωής ανθρώπων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εγκλήματα πολέμου. δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και φυσικά δεν συμφωνώ με το να διαμορφώσουμε ένα μηχανισμό που δήθεν θα νομιμοποιεί την άσκηση βίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας πρέπει να ανατίθονται ξεκάθαρα στις δημόσιες αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Συναδεινός. Κύριε Πρόεδρε, λόγω της αύξησης της τρομοκρατίας, του ασύμετρου των απειλών του τόπου και τρόπου τέλεσης τέτοιων ενεργειών, οι κρατικέ δυνάμει ασφαλεία αδυνατούν ω φαίνεται να ανταπεξέλθουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. το πλήθο και το εύρο των στόχων που υφίστανται στο δημόσιο και ιδιωτικό φάσμα μπορούν να ασφαλιστούν αποδοτικότερα με τη χρήση οργανωμένων εξοπλισμένων και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εταιρεών παροχή ιδιωτική ασφάλεια. αυτέ οι ιδιωτικέ εταιρείε θα μπορούν να συνεργάζονται εντό συγκεκριμένου πλαισίου με τι κρατικέ δυνάμει ασφαλεία σε επιχειρησιακό και πληροφοριακό επίπεδο απαιτείται όμως κατάλληλη διαμόρφωση της νομικής βάσης σαφής καθορισμός των κανόνων σύστασης και λειτουργίας τέτοιων εταιριών ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα υπέρβασης αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσίας αλλά κυρίως προβλήματα συνεργασίας και διαλειτουργικότητας που μπορεί να οδηγήσουν σε παράπλευρες απώλειες. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και η κυρία Μαρία Γραπίνη, το πέμπτο λεπτό του Κάτσι σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Μογκερίνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι υπέρ της έκθεσης ε, Φάουτμανς και είμαι υπέρ των συστάσεων που περιλαμβάνει η έκθεση. Γιατί έχουμε πια τα στατιστικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι εκατομμύρια πολίτες απασχολούνται σε αυτές τις, εταιρείες ιδιωτικής, τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Βέβαια δεν αντικαθιστούν το στρατό, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν περισσότερη ασφάλεια και άμυνα, οπότε είναι πολύ καλέ οι συστάσει υπέρ τέτοιων ε, ιδιωτικών ε, εταιριών ασφάλειας. Και την πράσινη βίβλο για του ενδιαφερόμενους. Και καλό είναι να έχουμε μια εναρμονισμένη στρατηγική για την πρόσληψη για στρατη, στρατιωτικούς σκοπούς τέτοιο, τέτοιου προσωπικού. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις εταιρείες αυτές με ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο κατακαιρματισμένη νομοθεσία και ρυθμίσεις για τέτοιες εταιρείες. Χρειαζόμαστε εναρμόνιση και σε νομικό και σε δικαστικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια οδηγία. Ευχαριστώ και ολοκληρώσαμε το πεντάλεπτο ΚΑΤΣΔΙ. Το λόγο έχει τώρα η πατή εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι χαιρετίζουμε την έκθεση που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις γνώσεις που έχουμε και στη συνειδητοποίηση αυτού του φαινομένου των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας που όπως είπατε μερικές φορές παίζουν κέριο ρόλο στην ασφάλεια και ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Και αυτή την άποψη ευθυγραμμιζόμαστε πλήρω με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή θεωρούμε ότι η πρόσληψη τέτοιων ιδιωτικών εταιριών είναι θεμητή νομότυπη, μπορεί να είναι και απαραίτητη και οι εταιρείε αυτές προστατεύουν και εργαζόμενους ε, στις ανθρωπιστικές ή άλλες οργανώσεις, αλλά φυσικά δεν ε, εξαιρούνται από το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αυτές οι εταιρείε και θα πρέπει να πληρούν τις ύψτες ε, προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει δυναμικό πλαίσιο, όπως μας επιθυμίζει η έκθεση, και οι ιδιωτικές εταιρείε ασφαλείας δεν λειτουργούν εν κενό, νομικό κενό και μάλιστα είμαστε η πρώτη ε, διεθνής οργάνωση που προσυπέγραψε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ε, που προώθησαν η Ελβετία και ο Ερυθρός Σταυρός για τη ρύθμιση των πρακτικών τέτοιων ιδιωτικών εταιριών. Θα πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε αυτό το πλαίσιο και να γίνει καθολικής εφαρμογή. Το Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών εξετάζει τη δυνατότητα διεθνούς πλαισίου για τη ρύθμιση και την εποπτεία τέτοιων ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας και ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει και να συμπληρώσει το Φόρουμ του Μόντρεαλ και την ε, οργάνωση για τον Διεθνή Διοντολογικό Κώδικα. Και είμαστε υπέρ της αναγνώρισης των αρχών του ΟΗΕ για, τε, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα αναγνωρίστηκε η αξία τους και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2016. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε λίγα σημεία. Καταρχήν, αν θέλουμε ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να επαφεθούμε στα κράτη-μέλη. Αυτά θα εξασφαλίσουν την πρόοδο και θα συμβάλλουν στην τροποποίηση των οδηγιών για τις κρατικές προμήθειες και των σχετικών κανόνων. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, όλοι οι πιθανοί ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν προσυπογράψει το Διεθνή Δοντολογικό Κώδικα και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ την εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων του Διδολογικού Κώδικα. Επίσης, ε, ε, το έργο αυτών των αναδόχων ε, προωθείται από τη χρήση μη επανδρομένων σκαφών και φυσικά θα πρέπει να επικαιροποιούμε το σύστημα ασφαλιστικών δικλείδων με τη συνεργασία επιστημόνων, πανεπιστημιακών, νόμομαθών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τι υπηρεσίες μπορούμε να αναθέτουμε εξωτερικά και τι θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των επαγγελματιών ε, στρατιωτικών δυνάμεων. Επίσης, συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Είχαμε στο δημόσιο τομέα πολλές τέτοιες εμπειρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον ιδιωτικό τομέα. Ε, μάλιστα τέτοιες ε, ιδιωτικέ ιδιωτικές συνεργάζονται πολλές φορές με το στρατό μας. Και καλό θα είναι να έχουμε την εκπλήρωση κοινών κανόνων και προτύπων με βάση τον Διεθνή Διοντολογικό Κώδικα. Πάνε δέκα χρόνια από τότε που άρχισε η κοινή γνώμη να ακούει για τέτοιε ιδιωτικέ εταιρείε. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι προ το συμφέρον όλων μα και προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συμβάλλουν οι εταιρείε αυτέ με το σωστό τρόπο στην εξασφάλιση τη ασφάλεια και του διπλωματικού μα προσωπικού και των απασχολουμένων στι ανθρωπιστικέ οργανώσει ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε για το συνεργάσιμο πνεύμα σας και ευχαριστώ που κι εσείς ε, επιταχύνατε τη συζήτηση και την ομιλία σας. Η ψηφοφορία της έκθεσης θα γίνει αύριο.